Καλημέρα σε όλους σας. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν την ε, εργασία μας, την ε, πρωινή μας συνεδρία. Έχουμε πολλές ψηφοφορίες σήμερα το πρωί. Πρώτον, σημείο 15. Να πω ότι κατεργήθηκε. Επομένως, δεν θα έχουμε ψηφοφορία επί του σημείου 15. Επίσης, Σημείο 16. Ψηφοφορία επί της διεθνούς εμπορικής πολιτικής στα πλαίσια των επιταγών της αλλαγής του κλίματος. Πρώτο συμβιβασμός υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 4. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 5 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 6 έχει ζητηθεί χωριστή ψηφοφορία. Ε, πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 7 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Φτάνουμε στο συμβιβασμό 2, ψηφοφορία κατά τμήματα, πρώτο τμήμα, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Συμβιβασμός 3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 μετρήσουμε λέει η Πρόεδρος ή μάλλον όχι, εγκρίνεται εγκρίνεται η 18 τροπολογία 19 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται προφορική τροπολογία Κυρία Πρόεδρε, το ΕΛΚ δεν δέχεται αυτή την προφορική τροπολογία.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 Σημείο 17. Τροποποίηση του κανονισμού υπηρεσιακή κατάσταση των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και του καθεστώτο που εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Τροπολογία 1. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 2. Υπέρ. Λοιπόν, ακούστε, υπάρχει ένα πρόβλημα, ένα λάθος στον κατάλογο ψηφοφορίας. Έχουμε δύο τροπολογίες στην, ε, επί της εκθέσεως Κασμάρεκα. Συμφωνείτε με τις δύο τροπολογίες αυτές, κύριε Κασμάρεκα. Ε, εγώ δεν τολμάω να ε, διαφωνήσω με τον κύριο Κασμάρεκα λέει ο κύριος Μίτσελ. Επομένως, ε, τροπολογία 2 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Να ψηφίσουμε λοιπόν επί της γνωμοδοτήσεως στο σύνολό της, έτσι όπως έχει τροποποιηθεί, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροποποίηση του κανονισμού του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση μηχανισμού χρηματοδότησης της αναπτυξιακής συνεργασίας. Επί της εκθέσεως ε, να σας πω ότι η τροπολογία 7 έχει αποσυρθεί. Τροπολογία 30 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβασμός 4 υπέρ κατά εγκρίνεται. Τροπολογία 32. Επί της 32 λοιπόν έχει ζητηθεί ψηφοφορία κατά τμήματα. Πρώτο τμήμα. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Όχι, καλύτερα να, καλύτερα να μετρήσουμε. Ξαναρχίζουμε. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κύριε Πρόεδρε, ενδεχομένω υπάρχει εδώ κάποια σύγχυση. Μιλάμε για την τροπολογία 32, δεύτερο τμήμα. Ακριβώς, το δεύτερο τμήμα της 32. Et donc c'était quoi On était où là Il était adossé, mais il faut Il faut le deuxième Alors c'est quoi Κοιτάξτε, υπάρχουν δύο τμήματα στο θέμα αυτό. Λοιπόν, είχαμε τρεις ψήφους υπέρ. Όχι, όχι. Συγγνώμη, λέει ο κ. Μίτσελ. Να ξαναψηφίσουμε το πρώτο τμήμα γιατί υπήρξε μία σύγχυση και νομίζω... Λοιπόν, μιλάμε για ψηφοφορία κατά τμήματα. Υπάρχουν τρία τμήματα όμως. Υπάρχει η ψηφοφορία η πρώτη και μετά η ψηφοφορία κατά τμήματα. Ψηφίζουμε την τροπολογία 32. Έχουμε ψηφοφορία κατά τμήματα που έχει ζητηθεί από τους σοσιαλιστές Πρώτο τμήμα. Κείμενο χωρίς ε, τις λέξεις από προξιμητέ μέχρι μέρ. Γυτνίαση με ιδιαίτερα περιφερειακές περιφέρειες ε, μέχρι τα υπερπόντια διαμερίσματα. Ακόμα υπάρχει σύγχυση. Λοιπόν, να ψηφίσουμε όμως ποιοι είναι υπέρ του κειμένου χωρίς το κείμενο που μόλις σας διάβασα από γυτνιάζουσα με περιοχές μέχρι υπερπόντια διαμερίσματα. Υπέρ. Κατά. Είχαμε 8 ψήφους υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Δεύτερο τμήμα. από προξιμητέ στο κείμενο στα γαλλικά μέχρι τη Ριτουάρ Ντουτρουμέρ, υπέρ κατά Εγκρίνεται. Τροπολογία 33 υπέρ κατά εγκρίνεται. Συμβιβασμός 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 35 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται προφορική τροπολογία του κυρίου Μίτσελ υπέρ κατά, αποχές, εγκρίνεται. Φτάνουμε στο συμβιβασμό 6 με ψηφοφορία κατά τμήματα. Πρώτο τμήμα, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Δεύτερο τμήμα, υπέρ, κατά απορρίπτεται. Τώρα πρέπει να ψηφίσουμε επί του συμβιβασμού 6. Ως έχει. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Donc, 37. 37. Υπέρ. Κυρία Πρόεδρε, νομίζω ότι πάλι έγινε ένα λαθάκι. Είχαμε δύο χωριστές ψηφοφορίες από αυτού. Ψηφίσαμε λοιπόν πρώτα τα δύο τμήματα και μετά ψηφίσαμε το συμβιβασμό. Εντάξει, μπορούμε να ψηφίσουμε, αλλά είχαμε τέσσερις ψήφους κατά. Θεωρώ λοιπόν ότι δεν, ε, ε, δεν πέρασε η, η χωριστή ψηφοφορία που, ζήτησε από τη, που ζητήθηκε από τους σοσιαλιστές. Α, έγινε και απερίφθη. Ψηφίσαμε και καταψηφίστηκαν τα δύο χωριστά τμήματα. Όχι, δεν κάναμε τέσσερις χωριστές ψηφοφορίες. Μια και υπάρχει σύγχυση, μήπως να ξαναρχίσουμε την ε, ψηφοφορία επομένως να ψηφίσουμε επί του συμβιβασμού έτσι όπως έχει τροποποιηθεί βάσει του αποτελέσματος των επιμέρους ψηφοφοριών ε, των κατά ψηφοφοριών. Monsieur Λυπούμε, λέει η Πρόεδρος, ο κύριος Γκέρεν. Κοιτάξτε, υπάρχει μια πρώτη χωριστή ψηφοφορία. Εκεί είχαμε αρνητική ψηφοφορία, αρνητικό αποτέλεσμα. Ε, και στη δεύτερη ψηφοφορία επίσης είχαμε αρνητικό και μετά έχουμε την ψήφο επί του συνόλου. Απερίφθη λοιπόν το πρώτο τμήμα, απερίφθηκε το άλλο και έχουμε τώρα την ψηφοφορία επί του συμβιβασμού δεν καταλαβαίνω γιατί έχει δημιουργηθεί το πρόβλημα αυτό και νομίζω ότι από συζήτηση στη συζήτηση θα δημιουργήσουμε πρόβλημα εκ του μειόντος και σύγχυση εκ της μειούσης. Πρόεδρος, θέλετε να διαβάσετε αυτό που ψηφίσαμε. κυρία Πρόεδρε. Νομίζω ότι δεν είναι απαραίτητο να ξαναδιαβάσουμε. Ψηφίσαμε τα δύο τμήματα βάσει του αιτήματο για χωριστή ψηφοφορία και μετά ψηφίσαμε επί του ε, συνόλου του, του συμβιβασμού έτσι όπως είχε τροποποιηθεί βάσει των προηγουμένων ψηφοφοριών. Επομένως, υπέρ του συμβιβασμού 6. Κατά. Αποχές Δεκτό ο συμβασμός 6. Donc, 11, Τροπολογία 11. Ποιος είναι υπέρ. Υπέρ, λέω. Κατά. Δεκτή. 38. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Η 12 έχει αποσυρθεί. Η 39 ψήφι υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. Η 13 έχει αποσυρθεί. 40 ψήφι υπέρ. Υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. 14 υπέρ. Κατά εποχές δεκτή. Μπορούμε να ψηφίσουμε όλες μαζί τις, τις ε, τροπολογίες το, της Επιτροπής Προϋπολογισμών 1 ως 5. Συμφωνείτε όλοι. Υπέρ, κατά, αποχές, δεκτές. Αιτιολογικές σκέψεις τώρα. Συμβιβαστική τροπολογία 1. Υπέρ, κατά, αποχές δεκτή. Τροπολογία υπερθμών 1, ψήφι υπέρ, κατά, αποχές δεκτή. 16 εκπίπτει, 17 υπέρ, κατά, αποχές δεκτή. Η 18 έχει εκπέσει. 21. Ψήφι υπέρ της 21. Αντίθετες. Πόσοι, τι. Υπέρ, επαναλαμβάνω λέει η πρόεδρος. Κατά. Απορρίπτεται λοιπόν. Συμβαστική τροπολογία παριθμών 2. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίθηκε. Συμβαστική τροπολογία 3. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Προφορική τροπολογία υπαριθμών 1. Υπέρ κατά αποχές δεκτή. Προφορική τροπολογία υπερθυμών 2 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Τροπολογία 29 υπέρ κατά αποχές απορρίπτηκε. Τροπολογία 28 ψήφι υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. Πέντε ψήφι υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. 6 υπέρ. Κατά. Α, αποχές εγκρίνεται και αυτή. Αιτιολογικές αναφορές, τροπολογία 15 ψήφι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Τελική ψηφοφορία. Η έκθεση όπως έχει τροποποιηθεί. Ψήφι υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Ομόφωνα. Θαυμάσιο. Πολύ ωραία. Μπράβο, μπράβο. Συγχαρητήρια κύριε Γκέρνς. Τώρα, ψηφίζουμε στο σημείο 19 της σημερινής διάταξης. Πρόκειται για τη θέση του Κοινοβουλίου για τον προϋπολογισμό του 2011. Έκθεση Μπέρμαν. είναι ανευτροπολογιών. Ψηφίζουμε λοιπόν τη γνωμοδότηση. Ψήφι ΠΕΡ. Κατά. τες εγκρίθηκε. Και τώρα και τώρα έχουμε τελειώσει τις ψηφοφορίες. Σας ευχαριστώ. Φυσικά συγχαίρω και τον εισηγητή, τον κύριο Μπέρμα, τον τελευταίο. Θα εξετάσουμε τώρα το σημείο 20 της ημέρας της διάταξης. Θα διακόψουμε για 5 λεπτά για να ξεκουραστούμε. Να ξελαχανιάσουμε, λέει η 5 λεπτά. στις 11 μείον 12. Nous reprenons notre Λοιπόν, προχωρούμε τώρα στη συζήτηση του σχεδίου γνωμοδότησης του κυρίου Μπάρτ και η γνωμοδότηση της Επιτροπής μας θα πάει στην Επιτροπή Εξωτερικού Εμπορίου που είναι η αρμόδια επί της ουσίας αφορά την απόφαση του Συμβουλίου σε σχέση με την εφαρμογή ορισμένων κατευθυντήριων γραμμών για τις εξαγωγικές πιστώσεις. Που έχουν, που έχουν ε, που έρχονται από δημόσια υποστήριξη. Και πρόκειται για την ε, συμπερίληψη της διάστασης ανάπτυξης, ώστε οι εξαγωγικές πιστώσεις να σέβονται τις ε, αρχές του αγώνα κατά της ένδυας και την συνεκτικότητα της πολιτικής ανάπτυξης. Κύριε Στάση, έχετε το λόγο λοιπόν. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, είχαμε συζητήσει το θέμα αυτό ήδη στην ε, ε, προηγούμενη μας ε, συνάντηση ε, αμέσως μετά από τις θερινές διακοπές και τώρα βρισκόμαστε σε μια φάση στην οποία πρέπει να εξετάσουμε και την ίδια την έκθεση και τώρα αυτό το οποίο μας ενδιαφέρει σε εμάς σε σχέση με τις ε, εγγυήσεις για τις εξαγωγικές πιστώσεις υπάρχουν φορείς οι οποίοι δίνουν τις εγγυήσεις αυτές σε όλα τα κράτη-μέλη και εδώ ο στόχος μας είναι να εξασφαλίσουμε ότι θα τηρηθούν οι κατευθυντήριες γραμμές. Είναι γραμμές κατευθυντήριες οι οποίες έχουν εγκριθεί στα πλαίσια μιας ε, εθελοντική συμφωνίας που θέλει τώρα το, η Κομισιόν να μεταβληθούν σε απόφαση της σύνολης Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Επιτροπή Οικονομικών Θεμάτων, η Επιτροπή Εξωτερικών Εμπορικών Θεμάτων είναι η αρμόδια για το θέμα αυτό. Και συνεργάστηκα πολύ καλά με τον ε, εισηγητή της Επιτροπής ΣΥΝΤΑ για σε επίπεδο νομοθετικό. Δεν είναι εύκολο να μετατραπεί μια εθελοντική Συμφωνία στα πλαίσια του ΟΟΣΑ και να τροποποιηθεί, να γίνει δεσμευτική. Πρόκειται για ένα μεγάλο σύνολο συμφωνιών και λεπτομεριών που καλύπτουν πάνω από 100 ε, σελίδες από ό,τι ξέρω. Ο εισηγητής επί της ουσίας και εγώ ο ίδιος είχαμε μεγάλες δυσκολίες για να μπορέσουμε να εξετάσουμε όλες αυτές τις παραγράφους και να δούμε πού χρειάζεται να υπάρξει μια τροποποίηση στις συμφωνίες του, του με συστηματικό τρόπο και από νομική έποψη νομίζω ότι κινούμαστε με τρόπο λίγο σκηνοτενή. Λοιπόν, είναι δύσκολο να είμαστε εξαντλητικοί στις τροπολογίες που θέλουμε να καταθέσουμε, γι' αυτό επιλέξαμε μια διαφορετική προσέγγιση βάσει της οποίας εξετάζουμε την οδηγία και προσπαθούμε να ενσωματώσουμε κάποιες από τις πτυχές που θεωρούμε ότι είναι απαραίτητο να συμπεριληφθούν σε αυτή Θέλουμε λοιπόν να εξασφαλίσουμε ότι θα μεταφερθούν όλα αυτά τα στοιχεία στην νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσα σε δύο παρατήματα. Καταρχήν έχουμε τη συμφωνία αυτή η οποία έχει γίνει στα πλαίσια του ΟΣΑ, αυτό είναι το ένα παράτημα και δεύτερον έχουμε ένα δεύτερο παράτημα που εξηγεί ποια ποιοι είναι οι δικοί μας στόχοι για τα αναπτυξιακά θέματα από την Επιτροπή μας. Έχουμε εν γέννη εννέα τροπολογίες τις οποίες έχω καταθέσει, οι πρώτες επτά από τις οποίες είναι καινοφανείς τροπολογίες, είναι νέες τροπολογίες σε ό,τι αφορά το κείμενο της οδηγίας και αφορούν τις αιτιολογικές σκέψεις. <clears throat> και έχουμε μόνο μία τροπολογία η οποία αφορά, για, αφορά τους στόχους της ε, νομοθεσίας και ενσωματώνει τους, ε, την συμφωνία του ΩΣΑ και αυτή αναφέρεται στο άρθρο 208 της Συνθήκης Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχει να κάνει με τα αναπτυξιακά θέματα και έχουμε επίσης την τροπολογία 9 που αφορά το δεύτερο παράδειγμα που υπάρχει μια πιο πλήρης απαρίθμηση του τρόπου με τον, τον ε, τρόπων με τους οποίους οι πιστοδοτικοί φορείς πρέπει να αντιμετωπίσουν τα θέματα αυτά. Και υπάρχει μια τροποποίηση που εγώ θέλω να επιφέρω στην εκθεσή μου και αυτό είναι κάτι που συζήτησα με την νομική υπηρεσία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Θα αποσύρω λοιπόν την τροπολογία μου υπαριθμών 9. Ελπίζω ότι το κείμενο αυτό έχει ήδη διανεμηθεί σε εσά. Έχω λοιπόν μια τροποποιημένη διατύπωση για την τροπολογία 9. Αυτή είναι μια τροπολογία λοιπόν που θα καταθέσω ως τροπολογία 9. Ποιος είναι ο στόχος λοιπόν όλων αυτών των μέτρων. Ο στόχος μας είναι για τις πρώτες 7 τροπολογίες οι οποίες προσθέτουν κείμενο στις αιτιολογικές σκέψεις, να αντιμετωπιστεί μια σειρά από θέματα τα οποία μας φαίνονται πολύ σημαντικά στην αναπτυξιακή πολιτική και κυρίως να εξασφαλίσουμε τη συνεκτικότητα μεταξύ των στόχων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην αναπτυξιακή πολιτική αφενός και αφετέρου τις δράσεις των πιστοδοτικών φορέων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι φορεί αυτοί φυσικά είναι αυτοί οι οποίοι χρηματοδοτούν τις αναπτυσσόμενες χώρες. Και αν δούμε τα αριθμητικά στοιχεία, περίπου 30 με 40% του χρέους των αναπτυσσόμενων χωρών έλκονται από αυτούς τους φορείς παροχής πιστώσεων. Είναι σημαντικές όλες αυτές οι ενέργειες ό,τι αφορά την εξωτερική βιομηχανία, τη δημιουργία υποδομών κτλ. Αλλά πρέπει όλοι αυτοί οι φορείς παροχής εγγυήσεων φαίνεται ότι έχουν άμεση σύνδεση με τα κράτη-μέλη πολλές φορές. Πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι η πολιτική που ακολουθούν αυτοί οι φορείς είναι η πολιτική την οποία θεσπίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Επομένως δεν ακολουθούν τη δική τους πορεία. Ότι δεν γίνονται δράσεις από αυτές οι οποίες αντιβαίνουν με την φιλοσοφία και την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης ό,τι αφορά την κλιματική αλλαγή, την, ε, τις κοινωνικές κτλ. Και φυσικά η κλιματική αλλαγή είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα μετά και από την θέση εφαρμογή της Συνδίκης Λισαβόνας. Θα σταθώ λίγα στις τροπολογίες αυτές για να σας εξηγήσω περί τίνος αναφέρομαι. Η τροπολογία 1 αναφέρεται στη, στα στη βαθμονόμηση των πτυχών του περιβάλλοντος και των κοινωνικών πτυχών που αρχίζουν πια να έχουν κάποια σημασία στο παγκόσμιο σύστημα επενδύσεων. Η τροπολογία 2 υπογραμμίζει το γεγονός ότι η υποστήριξη αυτών των φορέων στις αναπτυσσόμενες χώρες των πιστοδοτικών φορέων έχει γίνει μεγαλύτερη πηγή χρηματοδοτικής βοήθειας προς τις αναπτυσσόμενες χώρες και επομένως έχει κομβικό ρόλο Ίσως μπορώ να σας πω ότι τα σχέδια αυτών των πιστοδοτικών φορέων δίνουν έμφαση σε μεγάλες υποδομές όπως είναι παραδείγματος τα φράγματα, οι υποδομές εξορρυκτικού χαρακτήρα κτλ. Η τρίτη τροπολογία αναφέρεται στη συναντήση των G20 στο Pittsburgh και στο Τορόντο πέρσι και φέτος όπου οι G20 είχαν αποφασίσει ότι οι μη αποδοτικές επιδοτήσεις για ορυκτά καύσιμα θα πρέπει σταδιακά να καταργηθούν. Και τονίζω εδώ ότι οι κατευθυντήρες γραμμές του ΩΣΑ θα πρέπει να, ε, να συνάδουν με τα συμπεράσματα των G20. Η τροπολογία 4 τώρα κάνει σαφές ότι η μεταρρύθμιση των ε, ρυθμίσεων του ΩΣΑ θα πρέπει να έλθει σε πλήρη συμφωνία με το άρθρο 208 της Ευρωπαϊκής τη συνθήκη της ε, λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και εξηγώ λιγάκι τι αναφέρει το άρθρο 208. Πέμπτη τροπολογία τώρα. Αναφέρεται στο γεγονός ότι τα πρότυπα και οι αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να είναι κατευθυντήριες γραμμές στην παροχή βοήθειας από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αρχές για την προστασία του περιβάλλοντος, αρχές ανθρωπίνων δικαιωμάτων και όλες οι αρχές αυτές οι οποίες έχουν αποφασιστεί για τη δράση των επενδυτικών φορέων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπάρχει ένα εγχειρίδιο το οποίο λέει ακριβώ πρέπει να γίνει αυτή η χρηματοδότηση. Τροπολογία 6. Καλύπτει το, την ιδέα ότι οι προδιαγραφές σε επίπεδο περιβάλλοντος και κοινωνικού χαρακτήρα θα πρέπει να διατρέχουν όλο τον κύκλο των σχεδίων, όλη τη διάρκεια ζωής των σχεδίων για να εξασφαλίσουν την αηφορία τους και το να υπάρχει και εκτίμηση των κινδύνων για το περιβάλλον και τον κοινωνικό ιστό. Οποιοδήποτε σχέδιο των ε, φορέων αυτοχρηματοδότηση των ECA πρέπει να λαμβάνει αυτά υπόψη. Τροπολογία 7 αναφέρεται σε επίπεδα απόδοσης για το περιβάλλον και τον κοινωνικό χώρο που πρέπει να τηρούν αυτά τα σχέδια και αυτό συνδέεται με άλλες συμφωνίες που έχουμε για τις αϊφόρες πολιτικές, για την ε, συμφωνία της Κοτονού την ε, συμφωνία για την ε, ανάπτυξη και την συνοχή μεταξύ των δράσεών μας στην κλιματική αλλαγή. Μήπως πρέπει να μιλάω λίγο πιο αργά. Όχι. Η πρώτη χωρί μικρόφωνο. Ένα τέταρτο έχουμε μονάχα στη διάθεσή μας για να διεκπαιρεώσουμε αυτό το θέμα. Πρέπει να έχουμε και χρόνο για συζήτηση, αν μπορείτε να κλείσετε λιγάκι και να περιοριστείτε στα απαραίτητα. Τροπολογία 7, όπως σας είπα, αφορά τη σύνδεση με τις υπάρχουσες πολιτικές. Η τροπολογία 8 είναι λίγο ιδιαίτερη. Λέει ότι πέραν των συμφωνιών στα πλαίσια του ΩΣΑ, οι φορείς αυτοί, οι χρηματοδοτικοί φορείς, θα πρέπει να τηρούν αυτά τα οποία περιλαμβάνονται στο άρθρο 208 και η τροπολογία 9, η οποία είναι η μακροσκελέστερα. Αναφέρεται, έχει δύο τμήματα. Ο στόχος αυτής της τροπολογίας είναι να εξασφαλίσουμε ότι υπάρχει πλήρης διαβούλευση και διαφάνεια και πρόσβαση στην πληροφορία. Αυτό είναι το πρώτο τμήμα. Και το δεύτερο τμήμα αναφέρεται στις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθούνται από τους πιστοδοτικούς αυτούς φορείς ώστε να εξασφαλίστει και η συνοχή των δράσεών τους με τις κλιματικές αλλαγές μάλλον με την πολιτική μας στον τομέα της κλιματικής αλλαγής. Έχω διανύμει την τροποποιημένη μου τροπολογία. Ζητώ από τα μέλη της Επιτροπής να το εξετάσουν αυτό το έγγραφο και μπορούμε να επανέλθουμε με τους κοιόδης να δούμε αν πρέπει να κάνουμε κάποια αλλαγή και μπορώ να σταματήσω εδώ κυρία Πρόεδρε. Merci Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Βάνεν εδώ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έχετε το λόγο. Για δύο λεπτά. Ή κάποιος άλλος αν θέλει να πάρει το λόγο. Ναι, συγγνώμη. Πρέπει να πάρω το λόγο εκ μέρους του συναδέλφου. Άκουσα με ιδιαίτερο ενδιαφέρον ε, τον εισηγητή και ειδικότερα την, εξέταση των την ανάλυση των τροπολογιών. Πολλά, πολλές από τις απόψεις Ευρωπαϊκής ε, Επιτροπής καλύπτονται από τις ε, τροπολογίες σας και από τις κατευθυντήριες γραμμές. Εμείς μιλάμε κυρίως για τη μεταγραφή σε κοινοτική νομοθεσία του διακανονισμού. Οπότε... Πολλές από τις πτυχές ε, που αναφέρατε καλύπτονται από άλλες κατευθυντήριες ε, αρχές ε, του ΩΣΑ, αλλά και των, και των αποφάσεων που λήφθησαν στο Παρίσι από, τους, από την ομάδα των ε, πιστοδοτικών οργανισμών. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Σας υπενθυμίζω γιατί η προθεσμία για την υποβολή των τροπολογιών είναι η 3η 12 Οκτωβρίου το μεσημέρι, στις 12 το μεσημέρι και ότι θα ε, ψηφίσουμε στις 26 ε, Οκτωβρίου στην Επιτροπή μας. Περιμένουμε τώρα την κυρία Επίτροπο, η οποία θα έρθει από στιγμή σε στιγμή. Mm. Να μην διακόψουμε καλύτερα τις εργασίες μας. Έχω τη χαρά να καλωσορίσω μία ακόμη φορά την Επίτροπο Γεωργίευα, η οποία είναι πολύ πιστή στην Επιτροπή μας, έρχεται πολλές φορές να μας δει και στις 31 Αυγούστου είχε έρθει να μας δει για την ε, έκτακτη συνεδρίαση που είχαμε για την ανθρωπιστική βοήθεια στο Πακιστάν και σήμερα θα μας μιλήσει για το πρόγραμμα εργασίας της για το 2011. Κυρία Γεωργίευα, με πολύ μεγάλη χαρά σας δίνω το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Πρόεδρε, αξιότιμοι ευρωβουλευτέ, ε, κυρίε και κύριοι, αγαπητοί συνάδελφοι, χαίρομαι όλο ιδιαίτερω που βρίσκομαι και πάλι εδώ στην ε, Επιτροπή Ανάπτυξη ε, και με ενδιαφέρουν πάρα πολύ ε, αυτές ε, οι ε, συχνές συναντήσεις με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο γιατί εμπλουτίζουν τον προβληματισμό μου για τα βασικά θέματα της ανθρωπιστικής βοήθειας και πραγματικά αποτελούν τμήμα συνήθως της ημερήσιας διάταξής μου, του προγράμματός μας. Και τώρα θα μιλήσω αγγλικά. Σας ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρος λέει, μας εντυπωσιάσατε με τα γαλλικά σας. Μαθαίνω, μαθαίνω γαλλικά, λέει η κυρία Γεωργίευα. Και συνεχίζει στα αγγλικά. η στοχη μου είναι η εξή. Θα ήθελα καταρχά να σα ε, παρουσιάσω μία επισκόπηση του προγράμματο ε, τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το 2010. Για το ανθρωπιστικό κομμάτι θα σας πω κάποιες ιδέες για το 2011 και βεβαίως ε, θα σας παρουσιάσω εν γέννη το πρόγραμμά μου και στη συνέχεια θα περιμένω βεβαίως με ιδιαίτερη αγωνία τα σχόλιά σας και τη δική σας ε, καθοδήγηση. Θα ήθελα να ξεκινήσω με την εφαρμογή του προγράμματος για το 2010. Ήταν πραγματικά μία χρονιά με μεγάλες προκλήσεις, με μεγάλη ένταση, πολύ από, από πολύ απαιτητική χρονιά. Υπήρξαν πολλές ανθρωπιστικές ε, κρίσεις ε, σε πολλά μέρη του κόσμου και γι' αυτό ακριβώς μάλιστα φάνηκε ότι χρειαζόταν ε, το χαρτοφυλάκιο το οποίο ανέλαβα εγώ, την ανταπόκριση τη γρήγορη σε ανάγκες ανθρωπιστικέ βοήθειας. Χρειάστηκε πολλές φορές η υποστήριξή μας. Θα σας πω τα βασικά 10 προγράμματα IT, Πακιστάν, Σαχέλ, Σουδάν, Σομαλία, Μέση Ανατολή, Σρι Λάνκα, Κυργιστάν, Κολομβία και η περιοχή των μεγάλων λιμνών στην Αφρική. Και σίγουρα αφήνω πολλά απ' έξω πράγματα που δεν περιμέναμε, όπως για παράδειγμα ε, ο σεισμός στη Χιλή. Συνήθως ε, ε, δεν είναι χώρα η οποία λαμβάνει ανθρωπιστική βοήθεια η Χιλή. Θα ήθελα λοιπόν να αναφερθώ ειδικότερα ε, στην ΕΚΟ η οποία πραγματικά αντέδρασε πάρα πολύ γρήγορα στην ε, ε, διάθεση των ανθρωπιστικών πόρων και πρέπει να πω ότι γενικά ο μηχανισμός μας λειτουργήσε πάρα πολύ καλά, πολύ ομαλά, αποδοτικά και γρήγορα. Θα ήθελα επίσης να πω ότι ενώ από επιχειρησιακή απόψεως έγινε πολύ καλή δουλειά, ε, δούλεψαν πάρα πολύ σκληρά με την ομάδα μου επί των ε, προτάσεων πολιτικής ε, για, τα οποία, για τις οποίες θα επιμείνω. Το πρώτο βασικό ήταν το Μάρτιο, η πρώτη μου ανακοίνωση για την ανθρωπιστική βοήθεια για τα τρόφιμα, κάτι που ενέκρινε το Συμβούλιο και ήταν πάρα πολύ σημαντικό. Για δύο λόγους. Πρώτον, ε, όχι μόνο εισίδος δίνουμε ανθρωπιστική βοήθεια, αλλά προσπαθούμε να εστιάσουμε ε, την προσπάθειά μας και σε άλλους τρόπους ε, και σε τρόφιμα αλλά και σε παροχή ρευστού αν χρειάζεται ή άλλου είδους υποδομών κουπόνια για παράδειγμα γιατί πολλές φορές έτσι ενισχύεται και η τοπική ανάπτυξη και, καταλήγουμε και για να μην καταλήξουμε στην κατάσταση που έχουμε δει πολλές φορές, δηλαδή να δίνουμε εμεί τα τρόφιμα στον τοπικό πληθυσμό και τελικά ε, να σκοτώνουμε την τοπική οικονομία. Προσπαθήσαμε να το αποφύγουμε αυτό, ε, συνεργαστήκαμε πολύ καλά συνήθως με τους εταίρους μας, ακόμη και με εκείνους που ήταν κάπως πιο δικαστικοί, πιο διστακτικοί στο να αποφύγουν την εισίδος ε, βοήθεια τα τρόφιμα, δηλαδή απευθείας ανθρωπιστική βοήθεια υπό μορφή τροφίμων, ε, όπως για παράδειγμα ο Καναδάς διαφωνούσε με αυτήν την προσέγγιση. Όμως, καταλήξαμε τελικά στην ανάγκη επαναδιαπραγμάτευσης της Διεθνούς Σύμβασης για την Ανθρωπιστική Βοήθεια σε Τρόφιμα, γιατί δημιουργήθηκε τη δεκαετία του 60 και πρέπει να αναθεωρηθεί υπό το φως των εξελίξεων ε, των σημερινών. Τρεις βασικές πολιτικές ε, ήταν ε, οι πρωτοβουλίες μας, ε, οι οποίες ουσιαστικά θα είναι και η βάση των νομοθετικών προτάσεών μας για την επόμενη χρονιά. Δεν θα σας καταπλήξω αν σας πω ότι ένα βασικό σημείο είναι η ενίσχυση της άμεσης ανταπόκρισης. Έχουμε πάρα πολύ προχωρήσει στο θέμα αυτό, γιατί λαμβάνουμε υπόψη τα διδάγματά μα από τα τελευταία χρόνια και ειδικότερα από την ΑΕΤ και το Πακιστάν Φέτο. Ένας από τους βασικούς μας στόχους, ε, θα ήθελα όμως καταρχάς να πω, ότι ε, τα έχουμε καταφέρει πολύ καλά και μπορούμε να είμαστε πολύ ικανοποιημένοι από την ενίσχυση που ε, παρήχαμε, γιατί ήμασταν γρήγοροι και αποτελεσματικοί σε δύσκολες συνθήκες. Όμως μπορούμε να βελτιώσουμε ακόμη την κατάσταση και από εμά οι πολίτες περιμένουν να είμαστε σοβαροί, όχι μόνο να είμαστε γρήγοροι. Θέλουμε να βελτιώσουμε την συνέπεια, την ορατότητα της ανταπόκρισής μας στις κρίσης εντός και εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και γι' αυτό θα ήθελα να επιμείνω κυρίως στο βασικό θέμα. Αυτή τη στιγμή η ανάπτυξη των, της βοήθειάς μας βασίζεται σε επιτόπου ε, παροχή βοήθειας ε, και δεν έχουμε κανένα απολύτως ε, εναλλακτικό σενάριο για να μπορέσουμε να δούμε τι πόρους ακριβώς χρειαζόμαστε, για να μπορούμε δηλαδή να αναπτύξουμε αμέσως τους πόρους που θα χρειαστούν σε περίπτωση κρίσης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται ένα σύστημα που εξασφαλίζει ότι υπάρχουν βασικοί πόροι προς άμεση ανάπτυξη και ζητούμε από τα κράτη-μέλη να ε, να προβλέψουν εθελοντικά κάποιους, τέτοιου, κάποιους τέτοιους σπόρους για να μπορούμε να αντιποκριθούμε καλύτερα στην κρίση. Πρέπει επίσης ε, να υπάρχουν διακανονισμοί ε, για τις μεταφορές των πόρων σε περίπτωση ανάγκης ανθρωπιστικής βοήθειας. Αυτό είναι κάτι που θα μας επιτρέψει σε ε, έκτακτες περιπτώσεις, όπως με, για παράδειγμα θεομηνίες ε, μεγάλης κλίμακας, ε, να μπορούμε να αναπτύξουμε τους σπόρους μας μαζί και με στρατιωτικούς σπόρους αν χρειαστεί. Αυτά τα μέτρα θα είναι τμήμα των προτάσεων που τις ερχόμενες εβδομάδες ελπίζουμε μέχρι τα τέλη του Οκτωβρίου να έχουμε ολοκληρώσει την ανακοίνωσή μας και να σας την παρουσιάσουμε και να την παρουσιάσουμε προς έγκριση και στο Συμβούλιο. Είμαστε ιδιαίτερω ευγνώμονε ε, γιατί το Κοινοβούλιο μα ζήτησε πολλέ φορέ να είμαστε φιλόδοξοι στι προτάσει μα ε, και αναφέρομαι κυρίω στο σχέδιο έκθεση για τι νέε δυνατότητε άμεση ανταπόκριση, ε, μια έκθεση που την εξετάσατε χθε στην Επιτροπή σα. Περιμένω λοιπόν ε, εναγωνίω την αντίδραση του Κοινοβουλίου στην ανακοίνωση Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Επίση, θέλουμε να επεξεργαστούμε την ε, μεσοπρόθεσμη αναθεώρηση του σχεδίου δράση ανθρωπιστική βοήθεια. Ε, αναφέρεται η πρόοδο που έχει γίνει το 2007 από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη-μέλη. Εστιάζεται κυρίω στα πρακτικά αποτελέσματα στου έξι τομεί δράση ε, στους οποίους εστιάστηκε το ε, πρόγραμμα. Θα ήθελα να πω ότι η αναθεώρηση αυτή δεν είναι απλώς ένας τεχνικός απολογισμός. Δεν θέλουμε να εκλειφθεί έτσι, ειδικότερα επί τη βάση των προκλήσεων που αντιμετωπίσαμε αυτή τη χρονιά. Θέλουμε περισσότερη πολιτική ε, δυναμική στο πρόγραμμά μας, ε, γιατί ακριβώς οι κρίσεις που, που αντιμετωπίσαμε έδειξαν πόσο σημαντική είναι ε, η ύπαρξη ενός συνενετικού φιλόδοξου προγράμματος. Πρέπει να ενισχύσουμε τη μεγαλύτερη λογοδοσία για τα αποτελέσματα ε, της πολιτικής μας, ο κόσμος δεν ενδιαφέρεται τόσο πολύ για το πόσα λεφτά εξοικονομούμε. Ο κόσμος ενδιαφέρεται για το πόσες ζωές σώζουμε και πόσες ε, ανάγκες προσπαθούμε να εξυπηρετήσουμε. Και γι' αυτό ακριβώς πρέπει να εστιαστούμε και στην ορατότητα ε, υπ' αυτήν την έννοια του προγραμματός μας. Θέλουμε να είμαστε λοιπόν αποδοτικοί και αυτό είναι μια υψηλή προτεραιότητα και για μας και για τα κράτη-μέλη. Θέλουμε καλύτερη επίσης συνεργασία μεταξύ ε, άλλων εξωτερικών πολιτικών και της ανθρωπιστικής βοήθειας. Νομίζω ότι είναι κάτι που θα σας ενδιαφέρει και εσάς πολύ. Η συνεισφορά σας σε διεθνές επίπεδο λαμβάνεται σοβαρά υπόψη όχι μόνο από οικονομικής απόψεως, ε, αλλά πρέπει να ε, φαίνεται, να φαίνονται οι αξίες που υπερασπιζόμαστε σε διεθνές ε, επίπεδο. Εμείς ε, είμαστε σε συζήτηση με τα κράτη-μέλη για την προσπάθεια αυτήν ισχυμένης συνεργασίας και θα υπάρξει μέχρι το τέλος της χρονιάς ένα έγγραφο εργασίας σχετικά με το θέμα αυτό. Εμείς χαιρετίζουμε την ε, έκθεση της κυρίας Τρίφλερ για την ε, επί της ε, έκθεσης ιδίας πρωτοβουλίας μας έχει πραγματικά εντυπωσιάσει το έγκαιρο της εργασίας σας. Επίσης, το σώμα άμεσης ανταπόκρισης σε ανθρωπιστικές κρίσεις την ε, περασμένη εβδομάδα έγιναν οι διαβουλεύσεις με τους εμπλεκόμενους φορείς και πραγματικά με ενθάρρυνε όλος ιδιαίτερος η συζήτηση που έγινε γιατί επιτέλους δεν μου είπαν απλώ τι, τι δεν θα έπρεπε να γίνεται, αλλά μου είπαν τι θα έπρεπε να γίνεται. Δηλαδή ήταν πολύ πιο θετική η προσέγγιση και η προσέγγιση αυτή νομίζω ότι θα ενισχύσει πολύ περισσότερο τους στόχους και την, ε, από, την ε, επίτευξή τους. Αυτές ε, είναι οι τρεις βασικές μας προτεραιότητες και θα είναι και το βασικό, θα είναι το επίκεντρο ε, του προγράμματός μας για το 2011. Ο πρόεδρος Βαρόσο ε, ανέφερε ότι η αντιμετώπιση των καταστροφών ε, και η ανθρωπιστική βοήθεια είναι βασική μας προτεραιότητα και ότι θα είναι η βασικότερη νομοθετική πρόταση που θα υποβάλει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Όσον αφορά τα μέσα πολιτικής προστασίας, πρέπει να εφαρμοστούν οι συστάσεις που επεξεργαζόμαστε αυτή τη στιγμή και θα τονίσουμε ιδιαίτερα την ανάγκη αυτή. Όσον αφορά την μεσοπρόθεσμη αναθεώρηση, Πρόκειται για την αναθεώρηση της ε, σύμβασης του 96 η οποία πραγματικά μας βοήθησε πάρα πολύ, όμως πρέπει να την αναθεωρήσουμε για να δούμε ακριβώς υπό το φως των εξελίξεων ε, πώς ε, πρέπει να αναθεωρηθεί αυτός ο κανονισμός για την ανθρωπιστική βοήθεια. Η τρίτη νομοθετική ε, πρωτοβουλία θα αφορά ακριβώς το πλαίσιο της ανθρωπιστικής βοήθειας. Γιατί το επόμενο έτος θα είναι το έτος του εθελοντισμού. Θα έχουμε ένα πιλωτικό πρόγραμμα και παράλληλα θα επεξεργαζόμαστε την νομοθεσία που θα συμπεριλάβει τις εμπειρίες από το πιλωτικό αυτό πρόγραμμα. Οπότε το 2011 θα είναι ένα προπαρασκευαστικό έτος και το 2012 θα είναι το έτος της σχετικής νομοθετικής πρότασης. Όλες αυτές οι πρωτοβουλίες ε, πολιτικής δεν πρέπει να μας, ε, να μας παρεκκλίνουν από το βασικό μας στόχο που είναι η ανταπόκριση στις κρίσεις. Στην Παρασκευή αναφέραμε την, ε, στην ανάπτυξη της βοήθειας προς το Πακιστάν από 70 110 εκατομμύρια και περίπου 2 δισεκατομμύρια ανθρωπιστικής βοήθειας ε, για την ανάκαμψη. Επίσης ολοκληρώνουμε την επιχειρησιακή στρατηγική για το 2011 και στις αρχές του 2011 θα σας παρουσιάσουμε τις προτεραιότητές μας. Θα είναι βασική η προτεραιότητα ε, για το 2011 δηλαδή ετοιμότητα, ανταπόκριση, αποκατάσταση ε, και να μάθουμε από τις ε, από, το, από, από, το, από τις εμπειρίες μας ε, ως προς την αντιμετώπιση των κρίσεων. Μπορεί να μην είναι το βασικό ε, σημείο του προγραμματός μου, αλλά θα, είναι, ε, θα παραμείνει πολύ ψηλή μου προτεραιότητα. Θα ήθελα επίσης να ολοκληρώσω με μία παρατήρηση για την οικονομική πτυχή της ανθρωπιστικής ε, ενίσχυσης. Χρειάζεται περισσότερη ανθρωπιστική βοήθεια, όμως οι προϋπολογισμοί συνεχώς μειώνονται. Και Γι' αυτό πρέπει να προσπαθήσουμε να ε, χρησιμοποιήσουμε, να αξιοποιήσουμε με όσο το δυνατόν καλύτερο τρόπο το κάθε ευρώ που ξοδεύουμε. Και αυτό θα εξακολουθήσουμε να κάνουμε, σας διαβεβαιώ. Πρέπει όμως να αναγνωρίσουμε και το γεγονό ότι έχουμε ακολουθήσει τη μέθοδο να ε, ξοδεύουμε περισσότερα από όσα είχαν διατεθεί για την ανθρωπιστική βοήθεια. 1,1 δισεκατομμύρια ευρώ ήταν το κόστος φέτος. Ε, ήταν αυτά που τελικά εκταμιεύτηκαν με ένα προϋπολογισμό 800 εκατομμυρίων αρχικό. Έγιναν, σε σε, έγιναν όλα τα τελευταία 10 χρόνια με την εξαίρεση ενός έτους αυτό που σας λέω. Πρέπει λοιπόν να σας επιστήσω την προσοχή ότι υπάρχει έλλειψη πόρων για την ανθρωπιστική βοήθεια, για την πολιτική ε, προστασία. Ε, χρειαζόμαστε περισσότερους πόρους όταν, λένε, όταν μου λένε ότι χρειαζόμαστε περισσότερα χρήματα, απαντώ ότι όταν έχω όταν πηγαίνω σε μέρη όπου υπάρχουν ζητήματα ζωής ή θανάτου, εγώ είμαι υποχρεωμένη να διατηρήσω την ισχυρή ε, υποστήριξη των επιπλέον πόρων που χρειάστηκε κάθε φορά να διαθέσουμε και βέβαια θα είμαστε και πάρα πολύ απαιτητικοί ε, για τη λογοδοσία, ώστε να είστε περήφανοι για τα χρήματα που ξοδεύουμε. Σας ευχαριστούμε πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ. Κυρία Γκερέρο Σαλόμ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε. Πρώτα απ' όλα φυσικά θέλω να εκφράσω τις ευχαριστίες μου στην Επίτροπο για την παρουσία της στην Επιτροπή μας. Όπως αναφέρατε και εσείς είναι τακτική η παρουσία της και σίγουρα αυτό είναι κάτι το οποίο επενούμε ιδιαίτερα σαν μέλη της Επιτροπής αυτής το γεγονός ότι είναι διαθέσιμη και πάντα έτοιμη να εμφανιστεί ενώπιόν μας. Θέλω επίσης να συγχαρώ την κυρία Επίτροπο για το γεγονός ότι σε όλη τη διάρκεια αυτού του έτους, όπως τόνισε έτους το οποίο ήταν πυκνό σε ανθρωπιστικές καταστροφές. Για το γεγονός λοιπόν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση μπόρεσε να έχει μια σημαντική παρουσία για την αντιμετώπιση αυτών των καταστροφών και αυτό φυσικά οφείλεται σε μεγάλο βαθμό και στη δική σας θέληση να είσαστε παρούσα και να είσαστε κοντά στα προβλήματα των ανθρώπων που ανεφύησαν το 2010. Για το μέλλον τώρα, Πιστεύω ότι θα μπορούσαμε να φανταστούμε ότι οι ανθρωπιστικές καταστροφές, οι ανθρωπιστικές κρίσεις θα μπορούσαν να επαναληφθούν και με μεγαλύτερη ένταση στο μέλλον. Όχι για λόγους θρησκευτικού ή πολιτικούς, παρόν όχι επειδή έχω άμεση σύνδεση με τον Κύριο και μπορώ να προβλέψω ότι θα γίνει, αλλά γιατί η κλιματική αλλαγή θα έχει επιπτώσεις όλο και πιο έντονες σε διάφορα μέρη του κόσμου, όπως είδαμε φέτος ιδιαίτερα στο Πακιστάν και σε άλλες περιοχές του κόσμου, ιδίως της Ασίας. Όπως αναφέρατε λοιπόν κυρία Επίτροπε, χρειάζομαστε περισσότερα υλικά μέσα, περισσότερους πόρους, αλλά χρειαζόμαστε περαιτέρω και καλύτερο συντονισμό, ώστε να μπορέσουμε να επιτύχουμε δύο στόχους του οποίου αναφέρατε και εσεί στην παρέμβασή σα, Πρώτον, να έχουμε μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα και επίση για να έχουμε μεγαλύτερη ορατότητα. Και σχετικά, εγώ θα ήθελα να σα παροτρύνω και πιστεύω ότι και όλο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα υποστηρίξει μια τέτοια κίνηση να, για να υπάρχει μια, ένα στενότερο συντονισμό μεταξύ των ανθρωπιστικών φορέων των κρατών μελών και τον ανθρωπιστικό φορέα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις άλλες υπηρεσίες της Κομισιόν. Γνωρίζουμε ότι πολλές φορές υπάρχουν δισταγμοί και αντιστάσεις στα κράτη-μέλη, γιατί και οι φορείς τους θέλουν να διατηρήσουν την ορατότητά τους. Αλλά, όπως και σε άλλες πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πρέπει να τους πείσουμε ότι εάν είμαστε ορατοί σαν Ευρωπαϊκή Ένωση, όλα τα κράτη-μέλη είναι πιο ορατά από ό,τι μπορεί να είναι μεμονωμένα. Πρέπει να υπάρξει επίση μεγαλύτερο συντονισμό με τους διεθνείς φορείς κυρίως τι υπηρεσίες των Ηνωμένων και να βελτιώσουμε γενικά το συντονισμό σε διεθνές επίπεδο. Εσείς αναφέρατε το θέμα της προβλεψιμότητος που είναι ένας από τους στόχους στους οποίους θα πρέπει να επιζητούμε και να επιτύχουμε. Ένα από τα βασικά στοιχεία της προβλεψιμότητος όμως θα πρέπει να είναι και οι πόροι οι οποίοι εγγράφονται στον προϋπολογισμό. Εγώ ανέταμον τους προϋπολογισμούς των τελευταίων ετών, τον αρχικό προϋπολογισμό της Γενικής Διεύθυνσης Ανθρωπιστικών Θεμάτων ΕΚΟ, από το 2005 μέχρι το 2009 όχι μόνο είναι σταθεροί αυτοί οι προϋπολογισμοί αλλά μειώθηκαν ελαφρά. Αληθεύει όπως είπατε ότι τελικά μπορούμε να εξασφαλίσουμε πάντα πρόσθετους πόρους από άλλες γραμμές του προϋπολογισμού που έχουν σαν αποτέλεσμα σε τελική ανάλυση να διπλασιάζονται οι πόροι που πραγματικά εκταμιεύονται σε σχέση με αυτούς που προβλέπονται αρχικά στον προϋπολογισμό. Δεν είναι όμως η πιο πρόσφορη τεχνική προϋπολογισμού αυτή. Θα πρέπει να προσπαθήσουμε να αποφύγουμε το να γίνεται συνέχεια προσφυγή σε τέτοιες τεχνικές. Να ξέρουμε λοιπόν από την αρχή ότι χρειαζόμαστε ένα ορισμένο επίπεδο σε πόρους του προϋπολογισμού και όχι να βασιζόμαστε στο ότι όταν παρουσιαστούν προβλήματα θα μπορέσουμε να αποσπάσουμε κονδύλια από άλλες πηγές. Τέλος, θέλω να σας ζητήσω κάτι το οποίο φαίνεται ότι είναι μηχανιστικού χαρακτήρα, αλλά μπορεί να είναι χρήσιμο για τα μέλη της Επιτροπής μας. Ένα τμήμα λοιπόν της παρέμβασής σας, που να είναι κάπως πιο διευρυμένη η παρέμβασή σας σε επίπεδο τεκμηρίωσης, να μπορεί να αποστέλλεται στα μέλη της Επιτροπής μας για να έχουν καλύτερη γνώση των τεκτενομένων. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Φίσας. <clears throat> Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε για τις θαυμάσιες παρουσιάσεις σας αλλά και για τις δραστηριότητες που έχετε φέρει σε πέρας. Θέλω να κάνω κάποιες σκέψεις εδώ. Η πρώτη μου σκέψη είναι ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν κάποιες συγκρούσεις ή καταστάσεις έντασης για τις οποίες εμείς θα πρέπει να αναλάβουμε αμέσως ε, δράση Μιλήσαμε για την Αιτή, μιλήσαμε για το Πακιστάν φυσικά, αλλά εγώ θεωρώ ότι αυτές οι αναδυόμενες κρίσεις δεν πρέπει να μας κάνουν να ξεχάσουμε άλλες καταστάσεις οι οποίες βρίσκονται σε μια τελμάτωση εδώ και πολύ καιρό και δεν είναι στην πρώτη σελίδα των ε, εφημερίδων. Παραδείγματος χάρη η κατάσταση της Δυτικής Σαχάρας, των καταβλισμών των Σαχαραούι εκεί. Εκεί προφανώς ο άμεσος χαρακτήρας της ανάγκης δράσης στην ΑΕΤ στο Πακιστάν μπορεί να μας κάνει να παραγνωρίσουμε άλλες καταστάσεις οι οποίες χρονίζουν εδώ και πάρα πολλά χρόνια και δεν φαίνεται ότι είναι τόσο κατεπίγουσες αλλά είναι και αυτές καταστάσεις πολύ σημαντικές για τις οποίες θα πρέπει να αναλάβει δράση η Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα πρέπει να γνωρίζουμε ποια είναι η κατάσταση και ακόμα και όταν δεν είναι στα πρωτοσέλιδα ή στη στους κύριους τίτλους των καναλιών. Πάντα ξέρουμε ότι θα έρθουν και στο μέλλον άλλες τέτοιες έκτακτες καταστάσεις, αλλά αυτά δεν πρέπει να μας κάνουν να ξεχάσουμε καταστάσεις οι οποίες είναι σχεδόν μόνιμες. Επίσης, σε σχέση με το εθελοντικό σώμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μου φαίνεται αυτή η task force, αυτή η δύναμη κρούσης, η οποία αντιμετωπίσει τις καταστάσεις αυτές, θα πρέπει να έχει μεν εθελοντές, αλλά εάν δεν έχει τη σωστή πλαισίωση, μπορεί να είναι αναποτελεσματική η λειτουργία της. Δηλαδή, ήθελα να σας ρωτήσω αν έχετε κάποιες ιδέες σε σχέση με το πώς θα συγκροτηθεί αυτό το εθελοντικό σώμα. Κύριος Γκέρντς. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Όπως πάντα, με μεγάλη ικανοποίηση ακούσαμε για μια ακόμα φορά την κυρία Γεωργίεβα. Ε, δεν θα πω παραπάνω ε, όσον αφορά τα θετικά σημεία της εισήγησής της που είναι πολλαπλά. αλλά θέλω να αναφερθώ στην βραδύτητα ε, με την οποία ε, δίνεται η βοήθεια στο Πακιστάν. Ε, κοιτάξτε, εγώ δεν προσπαθώ απλώς να επιρρύψω ευθύνη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Περισσότερο στις πολύ πλούσιες χώρες της περιοχής. Πιστεύω ότι εκεί είναι μια καταστροφή φυσική, μια μεγάλη καταστροφή που θα έπρεπε πολύ γρήγορα να αντιμετωπιστεί. Ε, θα μπορούσατε να μας πείτε λοιπόν τι θα μπορούσε τουλάχιστον να, πει, να κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έτσι ώστε να πιέσει λίγο περισσότερο αυτές τις χώρες οι οποίες κρατούν ακόμα μια επιφυλακτική στάση. Ε, η περίπτωση αυτή είναι πολύ καλή όσον αφορά την ταχύτητα επέμβασης της, ε, Ευρωπα... της Ευρώπης. Όμως ε, θα ήθελα να αναφερθώ και σε κάποιους αριθμούς που με προβληματίζουν Νομίζω και το τονίζω, νομίζω ότι μπορώ να πω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ε, μακράν ο πρώτος ε, δωρητής όσον αφορά τις ε, πλημμύρες του Πακιστάν. Νομίζω λέω, γιατί δεν έχω συγκεκριμένα αριθμητικά στοιχεία. Πιστεύω ότι είναι πιο εύκολο στις μέρες μας ε, να, σε δεχτεί ο Πάπας ε, σε τέτα τέτ επίσκεψη παρά να έχεις πρόσβαση σε τέτοιου είδους αριθμητικά στοιχεία. Υπάρχει μια μεγάλη διάσταση ανάμεσα στην πραγματικότητα και την κατάσταση έτσι όπως περιγράφεται στις συνθήκες μας. Πότε θα μπορούσαμε να έχουμε έστω μία πρώτη, ένα πρώτο προσχέδιο ε, της ε, ε, κατάστασης όσον αφορά τις επεμβάσεις μας ε, και όσον αφορά τους προϋπολογισμούς μας. Κοιτάξτε, την εποχή που ζούμε όλο και πιο επιφυλακτική είναι η στάση των Ευρωπαίων φορολογουμένων και επομένως τουλάχιστον να πούμε σε αυτόν τον άνθρωπο που πληρώνει ότι ξέρεις κάτι κάναμε αυτά και αυτά. Ζήτησα λοιπόν κάποια αριθμητικά στοιχεία τα οποία έστω και στοιχειώδη και βασικά ήταν αυτά που ζήτησα παρόλα αυτά δεν μπορέσαν να μου τα δώσουν. Νομίζω λοιπόν ότι ε, θα πρέπει να δούμε ποιες είναι οι προσπάθειες που μπορεί να κάνει και ποιοι είναι οι πόροι που μπορεί να κινητοποιήσει κάθε χώρα μαζί με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεύτερον, με έκπληξη ε, διάβασα μία μελέτη, δεν θυμάμαι ακριβώς τον τίτλο της, που έλεγε, ασχολείται μάλλον με τον ευάλωτο χαρακτήρα ε, την ευάλωτη φύση των ε, ε, πτωχών χωρών απέναντι στις φυσικές καταστροφές. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα αλλάξει στρατηγική έτσι ώστε να ανταποκριθεί σε αυτήν την ιδιαιτερότητα γιατί φαίνεται ότι οι φυσικές καταστροφές μόνο θα αυξάνονται στο μέλλον και επομένως τι μπορεί να κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επ' αυτού. Γιατί ε, αν μπορούσατε να μου απαντήσετε ακόμα και σήμερα, αλλά έστω και αργότερα, εάν προτίθεστε να αλλάξετε λίγο τον γενικό σχεδιασμό. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Στίφλερ. Κυρία Επίτροπε, όπως πάντα είστε παρούσα έρχεστε σε επαφή μαζί σας, είστε παρούσα στις ε, συνεδριάσεις μας ε, και επομένως είναι εξαιρετική η στάση σας. Ε, είχα πολλές ερωτήσεις να σας κάνω, τις οποίες όμως απαντήσατε στην πρώτη σας παρέμβαση. Έχουμε πολλές επαφές με τη Γενική Διεύθυνση Ανθρωπιστικής Βοήθειας, την ΕΚΟ ε, νομίζω ότι πρέπει να κάνουμε μια ανάλυση όσον αφορά ε, ε, το συσχετισμό ανάμεσα στην ανθρωπιστική βοήθεια και τις οικονομικές δυσκολίες. Νομίζω λοιπόν ότι είναι σαφές ότι οι ανθρωπιστικές προκλήσεις μπορούν να απαντηθούν μονάχα μέσα από αυστηρή ε, συνένεση και αυστηρή εφαρμογή των σχεδίων δράσης αλλά θα πρέπει να έρθουμε σε επαφή και με όλους τους ανθρωπιστικούς παράγοντες ε, και να είναι ε, περισσότερο ορατή η συνένεση και να γνωστοποιείται και στα κράτη-μέλη. Επίσης Πρέπει να έχουμε πληροφορίες για τον τρόπο με τον οποίο τα κράτη-μέλη εφαρμόζουν, υλοποιούν αυτήν την συνένεση η ομάδα εργασίας του Συμβουλίου για την Ανθρωπιστική Βοήθεια θα μπορούσε να αποτελέσει το ε, ιδεώδες φόρουμ έτσι ώστε ε, να σιγουρευτούμε ότι γίνονται σεβαστές οι αρχές της συνένεσης. Ε, στη δεύτερη ερώτηση που ήθελα να θέσω απαντήσατε ήδη όσον αφορά τώρα την ορατότητα ευθυγραμμιστώ λίγο με τον κύριο Γκέρεντς. Ε, μιλάμε για τους ε, πολίτες μας και οι πολίτες ε, έχουν μόνο την αρνητική πληροφόρηση, η φυσική καταστροφή, τα πράγματα που δεν προχωράνε καλά, τι δεν πάει καλά και πολύ σπάνια μαθαίνουν τα θετικά πράγματα τα οποία έχουμε κάνει. Πώς είναι δυνατόν να περιμένουμε ότι θα εξακολουθήσουν να κινητοποιούνται οι πολίτες της Ευρώπης για τις μελλοντικές καταστροφές οι οποίες φεύ δεν μπορούν να αποφευχθούν. Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Γεωργίευα, μήπως μπορείτε να απαντήσετε στις ερωτήσεις αυτές. Ευχαριστώ πολύ για τις προτάσεις και τις ερωτήσεις ε, που μας ε, κάνατε. Επιτρέψτε μου να ξεκινήσω πρώτα ε, με την εκτίμηση ότι θα δούμε αύξηση και εντατικοποίηση των φυσικών καταστροφών λόγω των κλιματικών αλλαγών. Συμφωνώ με τη διαπίστωση αυτή. Ήδη από το 1975 έχουμε δει ότι έχουν πενταπλασιαστεί οι φυσικές ε, καταστροφές. Έχουν εξαπλασιαστεί, βλέπε, επταπλασιαστεί τα θύματα ε, και το οικονομικό κόστος των φυσικών αυτών καταστροφών. Βεβαίως ε, μπορούμε να κάνουμε μια σύγκριση και με την αύξηση της οικονομίας η οποία έχει αναπτυχθεί τρεις ή τέσσερις φορές από το 1975 ε, επομένως και σε σχέση με το ε, αεπ εάν πούμε ότι το αεπ είναι αυτό που εκφράζει την οικονομική ανάπτυξη τότε η οικονομική μας βάση αναπτύσσεται με βραδύτερο ρυθμό από ότι οι φυσικές καταστροφές και επομένως θα φτάσουμε κάποια στιγμή σε ένα κρίσιμο σημείο. Άρα χρειάζεται συντονισμός για πιο συντονισμένη αντίδραση. Σύμφωνο απολυτότατα με αυτήν την ε, θέση σας σχετικά με τον καλύτερο συντονισμό ε, μεταξύ μας και με τους άλλους έτσι ώστε να οργανώνουμε καλύτερα οποιαδήποτε μορφή ανθρωπιστικής βοήθειας νομίζω ότι θα πρέπει λίγο να ξεπεράσουμε και τα εσκαμμένα της παραδοσιακής μορφής ε, συντονισμού δηλαδή ανάλογα ε, με το είδος της φυσικής καταστροφής ε, θα πρέπει να έχουμε ένα ειδικό σενάριο αντιμετώπισης ποια, ποιοι είναι οι πόροι που χρειαζόμαστε, ποια είναι τα μέσα που χρειαζόμαστε έτσι ώστε να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε καλύτερα σε μια συγκεκριμένη φυσική καταστροφή, πώς μπορούμε να συντονιστούμε εμείς μεταξύ μας αλλά και με τα Ηνωμένα Έθνη. Ε, γι' αυτό έχουμε ξεκινήσει ε, και συζητήσεις ας πούμε με τους Αυστραλούς και τους Νέους Ζηλανδούς ε, για την περίπτωση των δασικών πυρκαγιών κυρίως γιατί όταν εμείς έχουμε χειμώνα εδώ εκείνοι έχουν καλοκαίρι και ανάποδα επομένως τα μέσα τα οποία έχουμε μπορούμε να τα διαθέτουμε ένα στον άλλον δεν είναι το σπουδαιότερο παράδειγμα ενδεχομένως, αλλά απλώς σας το λέω για να σας δείξω ότι θα πρέπει πολύ πιο συνολικά, πολύ πιο σφαιρικά να δούμε πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε και να ανταποκριθούμε σε τέτοιες φυσικές καταστροφές, να είμαστε πιο συντονισμένοι και πιο ορατοί. Θα απαντήσω, θα πάω αμέσως στο σχόλιο του κύριου Γκέρεν σχετικά με την ε, εικόνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όσον αφορά τα αριθμητικά στοιχήματα. Για το Πακιστάν, μπορώ να σας πω ότι μέχρι σήμερα έχουμε δεσμεύσει 400 ε, εκατομμύρια ε, ευρώ για ανθρωπιστική βοήθεια. 150 από την Ευρωπαϊκή ε, Επιτροπή. Μετά το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γερμανία και η Σουηδία είναι οι μεγαλύτεροι χορηγοί δωρητές. Δεν μπορώ να σας πω ακόμα ποιο θα είναι το τελικό συνολικό ε, αριθμητικό στοιχείο, αλλά να σας πω το εξής. Οποτεδήποτε μιλάω, μιλάω για την Ευρωπαϊκή Ένωση μέρος ε, της οποίας είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Όμως υπάρχει ένα ζήτημα. Το ζήτημα είναι ότι ε, οι ευρωπαϊκές χώρες είναι ευτυχείς όταν, ε, ε, όταν ε, μιλάει κάποιος εξ ονόματός τους, αλλά δεν είναι πάντα ευτυχής όταν πρέπει να συμβάλλουν με τον οβολό τους. Νομίζω ότι θα πρέπει να έχουμε ένα στοιχείο για την Ευρωπαϊκή Ένωση στο οποίο θα μπορούμε να συμβάλλουμε όλοι. Αυτός είναι ο καλύτερος δρόμος κατά την άποψή μου. Τουλάχιστον στον ανθρωπιστικό τομέα έτσι θα πρέπει να προχωρήσουμε. Ξέρετε, μερικές φορές μιλάω με τους συναδέλφους ε, στην ΕΚΟ ε, και συνήθως μιλάμε για τα δικά μας αριθματικά στοιχεία. Μου λένε λοιπόν ε, τόσα κάναμε στο Πακιστάν και αναφέρονται μονάχα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και δεν έχουν τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εγώ λέω πάρτε τα πίσω τα στοιχεία αυτά γιατί θέλω να έχουμε συνολικούς αριθμούς. Σχετικά με την προβλεψιμότητα των πόρων κατανοώ ότι έχει δημιουργηθεί ένα ικανό αποθεματικό αλλά ήταν καλό για 10 χρόνια πριν, αλλά έχουν αλλάξει οι συνθήκες, ο κόσμος έχει αλλάξει και πλέον όλα τα αποθεματικά αυτά ε, ενσωματώνονται στο προπολογισμό, επομένως δεν έχουμε, ε, δεν έχουμε το, το απαραίτητο ε, απόθεμα. Θα πρέπει να, δούμε, να βρούμε με τρόπους δημιουργικούς πώς θα κινητοποιήσουμε πόρους. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, αν κάθε χρόνο βλέπουμε ότι χρειαζόμαστε ένα δι για τέτοιου είδου παρεμβάσει, γιατί δεν βάζουμε από την αρχή στον προπολογισμό αυτό το ένα ε, δις. Ναι, βεβαίως ε, διανύουμε περιόδους ε, κρίσης that is baseline, in... και λιτότητας, αλλά 97% του κόσμου θέλουν να συνεχίσουμε αυτήν την ανθρωπιστική βοήθεια. Εγώ περιμένω λοιπόν ε, να δει κάποιος και να πει αντικειμενικά ότι ορίστε κάθε χρόνο, κάθε χρόνο ξοδεύουμε ένα εκατομμύριο και πλέον ε, και επομένως ε, θα πρέπει να μπουν στον προϋπολογισμό αυτά. Ξέρετε, δίνουμε πάνω από ένα δις και πάντα βρισκόμαστε αντιμέτωποι με πάρα πολύ δύσκολες επιλογές. Διαρκώς πρέπει να κάνουμε δύσκολες επιλογές. Και πιστεύω ότι θα πρέπει να έχουμε λοιπόν ε, και έχετε πάρα πολύ δίκιο ότι όταν φεύγουν οι προβολείς πάνω από ένα θέμα δεν μπορούμε να αφήνουμε τον κόσμο να πεθαίνει. Δεν έπεται ότι επειδή ένα ζήτημα έχει φύγει από το φως της δημοσιότητας δεν πρέπει να κάνουμε τίποτα για αυτούς. Ε, για τους πρόσφυγες ας πούμε, εδώ και 35 χρόνια έχουμε για του Σαχαράουι που είπατε ε, υπάρχουν ακόμα τέσσερα στρατόπεδα με πάρα πολύ κόσμο. Εδώ και 35 χρόνια είναι τα, τα στρατόπεδα αυτά και δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Δεν έχουμε κάνει κάτι για αυτούς. Δυσκολευόμαστε ε, για τον καθαρισμό του αριθμού τους. Δεν ξέρουμε. Λέμε ότι είναι 90.000 ε, οι ευάλωτοι ε, πληθυσμοί, αλλά δεν είμαστε σίγουροι. Στηρίζουμε ε, στηρίζουμε ε, την, ε, την περίπτωση αυτή αλλά βεβαίως δεν είναι ικανοποιητική, δεν είναι αρκετή. Αλλά τουλάχιστον τους ανακουφίζει κάπως. Έτσι ώστε να ανταποκριθούν στις πολύ βασικές τους ανάγκες. Νομίζω ότι παντού πρέπει να υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Αλλά δεν είναι δυνατόν για τα επόμενα ακόμα 35 χρόνια να αγνοούμε το πρόβλημά τους. Θα πρέπει να βρεθεί και κάποια πολιτική λύση. Και σε αυτή την περίπτωση αλλά και σε άλλες περιπτώσεις δεν θα ξεχάσουμε ε, τις ξεχασμένες κρίσεις δεν θα αφήσουμε τον κόσμο να πεθάνει επειδή ε, από τα, από τα πρωτοσέλιδα Ε, και βεβαίως μπορούμε να σας δώσουμε και περαιτέρω πληροφορίες για το θέμα αυτό όσον αφορά το εθελοντικό σώμα. Μέχρι τώρα έχουμε συμφωνήσει με τα υπόλοιπα ενδιαφερόμενα μέρη ότι θα έχουμε τρία στοιχεία δηλαδή ε, όσον αφορά αυτό το εθελοντικό σώμα και θα δούμε τι μπορούμε να κάνουμε με το νέο αυτό σώμα στους τρεις τομείς δηλαδή στην ε, ε, εξέβρεση ας του προσωπικού, στην εκπαίδευση και στην χρήση του. Και βεβαίως να μην εργαστούμε μόνοι μας, αλλά σε συνεργασία με εθελοντικές οργανώσεις για να δούμε πώς μπορούμε να καλύψουμε κάποιους νέους τομείς. Ας πούμε, προετοιμασία προς αποφυγή φυσικών καταστροφών ε, με ε, φύτεμα δέντρων, ας πούμε, έτσι ώστε να ενισχύσουμε τα δάση της ε, κάποιας περιοχής. Να δουλέψουμε λοιπόν μαζί με εθελοντικές οργανώσεις έτσι ώστε να καθορίσουμε κάποια πυρηνικά στοιχεία τα οποία θα είναι σημαντικά. Τώρα, αυτό το σώμα ε, θα ενταχθεί στο ήδη υπάρχον ε, εθελοντικό σχήμα το οποίο έχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή θα ενταχθεί στο δυναμικό της ΕΚΟ όλα αυτά αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης και ε, διαβούλευσης. Εντάξει, θα, θα, θα κάνουμε το πολιτικό πρόγραμμα, θα το εφαρμόσουμε, θα δούμε πριν την και μετά θα έρθουμε μια νομοθετική πρόταση ενώπιόν σας. Αυτό το οποίο είπε ο κύριος Γκέρενς προηγουμένω για τις φτωχές χώρες, τις χώρες που έχουν ευάλωτες δομές, είναι γεγονός. Η ζωή δεν είναι δίκαια αυτοί οι οποίοι έχουν συμβάλει περισσότερο στην αλλαγή πολλές φορές είναι αυτοί οι οποίοι πλήττονται περισσότερο. Και γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό να έχουμε δομές για τη μείωση του κινδύνου και την αντιμετώπιση των κρίσεων μέσα στην αναπτυξιακή με στρατηγική. Εγώ πηγαίνω στι αιτήσει συναντήσει του παλιού μου εργοδότη, τη Παγκόσμια Τράπεζα και του Διεθνού Νομισματικού Ταμείου για να μπορέσουμε να έχουμε μια κοινή στάση με του παγκόσμιου αυτού φορεί για να ενισχύσουμε τι δομέ και την ανθεκτικότητα των φτωχών χωρών έναντι του κινδύνου κυρίω τη κλιματική αλλαγή. Όχι μόνο τη κλιματική αλλαγή, υπάρχουν άλλοι παράγοντε, δημογραφική αστικοποίηση σε πτωχέ χώρε. Δεν ξέρω πόσοι από εσά έχετε πάει σε πραγματικά φτωχέ χώρε, σε αστικούς, αστικές συγκεντρώσει φτωχών χωρών. Είναι τεράστιες οι προκλήσεις. Πολλές φορές αυτά γίνονται με οικοδόμηση σε περιοχές όπου δεν θα έπρεπε να ζουν άνθρωποι. Τόσοι άνθρωποι πέθαναν γιατί είχαν χτίσει τα σπίτια του εκεί που δεν θα έπρεπε να είναι τα σπίτια. Είναι ένα σημαντικό θέμα και θα είμαι ειλικρινή μαζί σα. Δεν έχουμε προχωρήσει αρκετά στο θέμα αυτό. Οι εκπρόσωποι τη ΕΚΟ που είναι εδώ μπορούν να σα το εξηγήσουν, να σα το επιβεβαιώσουν. Έχουμε ένα μεγάλο πρόβλημα για να βοηθήσουμε τι ε, κοινότητε αυτέ τι τοπικέ να μειώσουν τι επιπτώσει των φυσικών καταστροφών. Πρέπει να κάνουμε περισσότερο όμως στον τομέα αυτό της μείωσης των κινδύνων καταστροφών. Και αυτό στη συνεργασία με τους συναδέλφους μας της ανάπτυξης. Γιατί όσο πιο ευάλωτες είναι αυτές οι κοινότητες, τόσο πιο πολλά άτομα θίγονται από τις αυτοπιστικές κρίσεις. Ό,τι μπορούμε να κάνουμε λοιπόν για να υπάρχει καλύτερη εκπαίδευση στον τομέα αυτό θα είναι θετικό. Και απαντάω σε αυτά που είπε η κυρία Στρίφλερ για το να γίνει πιο σαφές το μήνυμά μας. Ένα από τα προβλήματά μας είναι ότι έχουμε πολλές φορές να κηρύττουμε σε αυτούς οι οποίοι ήδη έχουν ασπαστεί τη θρησκεία μας. Τα λέμε αυτά τα πράγματα μεταξύ μας, βγαίνουμε από την αίθουσα και δεν γίνεται απολύτως τίποτα. Είναι ένα πρόβλημα ότι μιλάμε για μία συνένεση η οποία υπάρχει όμως μονάχα στην κοινότητα που ασχολείται με τα ανθρωπιστικά θέματα. Αλλά αυτή η συνένεση δεν έχει μεταλαμβανθευτεί και σε άλλους τομείς, σε άλλους χώρους όπως θα έπρεπε και το ίδιο με την ιδέα της μείωσης των κινδύνων καταστροφών. Συμφωνώ λοιπόν με την κυρία Στρίφλερ ότι υπάρχει ένας πολύ σημαντικός ε, ρόλος για μας να μπορέσουμε να έχουμε μια μεγαλύτερη απήχηση. Ήμουνα πρόσφατα στην ε, ε, Βασιλική Στρατιωτική Ακαδημία του Βελγίου και μίλησα μαζί τους για τα θέματα συνεργασίας πολιτικής και στρατιωτικής δράσης για την ανθρωπιστική ανακούφιση. Είναι σημαντικό λοιπόν να μπορούμε να έχουμε την απαραίτητη απήχηση στους χώρους εξουσίας κάθε φορά που αυτό είναι απαραίτητο. Τρεις. Κύριε Αγγέλος, και στο Πακιστάν λοιπόν ήμασταν παρόντες, έπρεπε να πω. Δεν καθυστερήσαμε, δεν χρονοτριβήσαμε. Ίσως δεν πέρασε αυτό στα μέσα ενημέρωσης, αλλά στις 31 Ιουλίου η Κομισιόν ήταν η πρώτη η οποία έδωσε κατευθείαν 30 εκατομμύρια ευρώ μια σημαντική βοήθεια και μετά αυξήσαμε αυτή τη βοήθεια, αλλά σίγουρα δεν έγινε γνωστό αυτό και συζητώ συγγνώμη για αυτό τώρα που παρενέβη. Κύριε Ασέν, έχετε το λόγο. Ε, ε, σας ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, χαίρομαι πολύ που σας καλωσορίζω σε αυτή την Επιτροπή και μετά τη συζήτηση που είχαμε και στην Επιτροπή Περιβάλλοντος επίσης. Θέλω καταρχήν να εκφράσω την υποστήριξή μου για την κατεύθυνση που ακολουθούν οι προτάσεις σας. και καταρχήν για την πρόληψη των ανθρωπιστικών κρίσεων και για την εστίαση που έχετε στο να μπορέσει να υπάρχει μεγαλύτερη ανθεκτικότητα των τοπικών κοινωνιών. Σύμφωνο λοιπόν με όλες αυτές τις προτάσεις που έχετε διατυπώσει, όπως είπατε, όσο και να είναι κανείς συντηρητικός σε δημοσιονομικό επίπεδο, η πραγματικότητα μας υποχρεώνει να αναζητήσουμε και περισσότερες πηγές χρηματοδότησης για να αντιμετωπίσουμε όχι μοναχά αναπτυξιακά προβλήματα, αλλά και τις ανθρωπιστικές κρίσεις στη διάσκεψη κορφής του ΟΗΕ επανελήφθη η πρόταση αυτή να υπάρξει ο φόρος χρηματοοικονομικών συναλλαγών. Αυτή τη φορά αυτή η πρόταση υπευλήθηκε πάλι από την ομάδα για καινοτόμε λύσεις για να αντιμετωπιστούν τα αναπτυξιακά θέματα. Το έχει επίσης τονίσει αυτό και το Κοινοβούλιο την ανάγκη τέτοιου φόρου και είπε και το Συμβούλιο ότι αν σε παγκόσμιο επίπεδο εγκριθεί μια τέτοια ιδέα για φόρο χρηματοοικονομικών συναλλαγών θα το υποστηρίξει και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Λόγω της αντίδρασης του Καναδά και άλλων χωρών δεν καρποφόρησε αυτή η προσπάθεια, αλλά ο πρόεδρος Μπαρόζου είπε ότι είναι έτοιμος να συζητήσει κάτι σχετικό. Αλλά, όπως μας είπε σε μια συνάντηση που είχαμε κατά τη διάρκεια της διάσκεψης κορυφής του ΟΗΕ για τα αναπτύξιακά θέματα, θα ήταν πολύ <clears throat> δύσκολο να διοχετευτούν τα χρήματα τα οποία προέρχονται από αυτό το φόρο στις ανάγκες ανάπτυξης που πρέπει να εξυπηρετήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα ήθελα λοιπόν να έχω και την άποψή σας για αυτό το θέμα. Υποστηρίζετε την ιδέα αυτού του φόρου. Είναι κάτι το οποίο βάσει των ε, πραγματικότητων που αντιμετωπίζεται είναι ένας φόρος ο οποίος θα ήταν απαραίτητο να εφαρμοστεί και αν υπάρξει ένας τέτοιος φόρος δεν θα πρέπει ένα σημαντικό τμήμα αυτού του φόρου των προσόδων αυτού του φόρου να χρησιμοποιείται για την ε, ανάπτυξη και την ε, ανθεκτικότητα στις κλιματικές αλλαγές. Ευχαριστώ. Ο κύριος Νιούτον Ντάν. Κυρία Επίτροπε, θέλω να κάνω δύο παρατηρήσεις. Μιλήσατε για την ανάγκη λογοδοσίας. Πολύ καλά. και ο κ. Σασένς και εγώ ήμασταν στην αντιπροσωπεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για, την, ε, για τους στόχους της ε, χιλιετίας και είδαμε ότι ορισμένε από τα αφρικανικές χώρες δεν θέλαν το έγγραφο αυτό του ΟΗΕ να αναφέρεται στην ανάγκη λογοδοσίας. Αυτό μας σοκάρισε. Και εσείς και εμείς ενδιαφερόμαστε πάρα πολύ για το θέμα αυτό του να είναι υπόλογες οι αρχές. Αλλά Κάτι το οποίο μας ενδιαφέρει είναι να τονίσουμε ότι οι πολίτες μας αυτή τη στιγμή στενάζουν κάτω από τις μειώσεις του προϋπολογισμού και των δημοσίων δαπανών που έχουν επιβληθεί λόγω κρίσης και θα πρέπει να κάνετε σαφές ότι και εμείς ως Επιτροπή Αναπτύξεως του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου πιέζουμε και εμείς για λογοδοσία και δεν είσαστε μόνο εσείς που το ζητάτε. Το άλλο θέμα που ήθελα να δείξω είναι το εξής μήπως μπορείτε να μου περιγράψετε το εξής, όταν υπάρχει μια κρίση που ξεκινάει στο Πακιστάν ή στην Αϊτή και λένε όλα τα κράτη-μέλη ότι ναι, ναι, θα συμβάλλουμε, υπάρχει κάποιος συντονισμός. Λέει δηλαδή μια κυβέρνηση, εμεί θα δώσουμε κουβέρτες, η άλλη λέει θα στείλουμε φάρμακα, θα στείλουμε σκηνές. Υπάρχει συντονισμός ή η κάθε μία κυβέρνηση δίνει τα δικά της δώρα και δίνουν όλοι παραγωγός τρόφιμα και καθόλου φάρμακα. Υπάρχει τρόπος να εξασφαλίσετε ένα συντονισμό ε, των, δωρεών που γίνονται. Η κυρία Κρέτου. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Και εγώ θα ήθελα να σας ευχαριστήσω κυρία Επίτροπε για την ενεργητικότητά σας και αυτό φάνηκε και στην ε, συνάντηση που είχαμε στο Στρασβούργο όταν τόνισα με, ε, ότι για το θέμα του Πακιστάν ήταν απόλυτα ικανοποιητική δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όπως είπατε και εσείς, πρέπει να δίνουμε περισσότερα μηνύματα προς τους διεθνείς φορείς ενημέρωσης και να εξηγήσουμε κιόλας και ότι λόγω της μεγάλης διαφθοράς που σοβεί στο Πακιστάν πολλά από τα εγχειρήματά μας, πολλές από τις προσπάθειές μας δεν μπόρεσαν να να φέρουν τη βοήθεια στους πραγματικούς αποδέκτες. Αυτό έχει να κάνει με τις δομές του ίδιου Πακιστάν. Και ήθελα να σα θέσω αυτό το ερώτημα. Σε ποιο βαθμό εσεί μπορείτε να εξασφαλίσετε ότι τα ποσά τα οποία εμεί αποφασίζουμε πραγματικά φτάνουν στα θύματα των φυσικών καταστροφών. Πώ μπορείτε να εξασφαλίσετε λοιπόν ότι τα χρήματα αυτά πιάνουν τόπο και σε ό,τι αφορά την ευρωπαϊκή, ευρωπαϊκή ανακουφιστική βοήθεια νομίζω ότι υπάρχει και ένα παραπάνω πρόβλημα. Η εξασφάλιση της ακεραιότητας και της ασφάλειας αυτών οι οποίοι παραδίδουν αυτή τη βοήθεια εκεί. Υπάρχουν πάνω από 100 άτομα τα οποία βρέθηκαν σε κίνδυνο κατά τη διάρκεια της ε, προσπάθειάς τους να παραδώσουν την ανθρωπιστική βοήθεια και θα ήθελα να ρωτήσω ακριβώς πώς μπορούμε να εξασφαλίσουμε την ασφάλεια αυτών των ανθρώπων που μπορεί να παίξουν και τη ζωή τους κοροναγράμματα για να παραδώσουν αυτή τη βοήθεια. Τέλος, θα ήθελα να σταθώ στο θέμα της δυνατότητας ταχείας αντίδρασης για την ε, αντιμετώπιση των κρίσεων, δηλαδή αυτής της ειδική μονάδας η οποία λειτουργεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θέλω να σας ευχαριστήσω εσάς προσεκτικά, προσωπικά μάλλον, για το γεγονός ότι όταν η Ρουμανία επλήγει από φυσικές καταστροφές επισκεφτήκατε τη χώρα μου. Ξέρω ότι τα εργαλεία τα οποία έχουμε για να μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε τους πόρους μας για την αντιμετώπιση των φυσικών καταστροφών μπορούν να απελευθερωθούν μόνο κατά προποθέσει. προϋποθέσεις. Και γι' αυτό πιστεύω ότι πρέπει βέβαια να σεβόμαστε αυτές τις προδιαγραφές, αλλά είναι και παράδοξο το ότι για το Πακιστάν παραδείγματος χάρη χρειάστηκε να περιμένουμε τρεις μήνες για να μπορέσουμε να κινητοποιήσουμε αυτά τα κονδύλια, ενώ για την ΑΕΤ αυτό έγινε από τη μια μέρα στην άλλη. Μήπως λοιπόν μπορεί να υπάρξει ένας τρόπος βελτίωσης και τροποποίησης του νομοθετικού πλαισίου, ώστε και στι καταστροφές που λαμβάνουν χώρα στην Ευρώπη να μπορεί να υπάρξει μια ταχεία απόκριση από αυτήν την ομάδα την ειδική που υπάρχει για την αντιμετώπιση κρίσεων. Όλα αυτά ήταν πάρα πολύ ενδιαφέροντα. Και βέβαια δεν ήταν και εύκολα. Όσον αφορά τον φόρο για τις ε, χρηματοοικονομικές συναλλαγές. Ναι, <coughs> είναι βέβαια ε, δυνατόν ε, να προκύψουν έσοδα με την εισαγωγή ενός ε, τέτοιου είδους φόρου χρηματοοικονομικών συναλλαγών. Δεν ξέρω πώς ακριβώς να απαντήσω, γιατί ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να το κάνουμε. Ο ε, χρηματοοικονομικός τομέας είναι ένας τομέας ε, που δεν φορολογείται ε, πολύ. Βέβαια είναι και ψηλή και μεγάλη κίνδυνη, αλλά το κατά πόσο εμεί θα έπρεπε να πληρώνουμε ω πολίτε τέτοιου είδου φόρο για, ε, ε, για το δημόσιο καλό, εντάξει, ναι μεν είναι καλή ιδέα, αλλά πρέπει να είναι παγκόσμιο κάτι τέτοιο για να έχει νόημα. Να δούμε τι θα γίνει στον επόμενο γύρο διαπραγματεύσεων. Για την ώρα είναι ευνοϊκό το περιβάλλον, ε, γιατί σε παγκόσμιο επίπεδο οι πολίτες είναι τόσο αποχοητευμένοι, όχι μόνο με, το, με την κρίση, αλλά ε, και με την κακή συμπεριφορά του οικονομικού τομέα, για να το πω έτσι. είναι η πρώτη δυσκολία. Το, η άλλη δυσκολία είναι να συμφωνήσουν όλοι, οι Ηνωμένε Πολιτείε, Κίνα, όλοι από αυτού. Ναι, μπορούμε να το κάνουμε όπως κάναμε και με το πρόγραμμα εμπορίας ε, αερίων. Τα καταφέραμε αρκετά καλά Βέβαια είμαστε και 500 εκατομμύρια. Είναι, είναι δυνατόν να λειτουργήσει ένα τέτοιο σύστημα σε ευρωπαϊκό επίπεδο μόνο όμω ε, για τον ε, φόρο τον οποίο αναφέρατε δεν ξέρω κατά πόσο ε, έχει νόημα να το κάνουμε μόνο σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Επίσης, εντάξει, από ό,τι κατάλαβα υπάρχει διάθεση να κάνουμε μια τέτοια προσπάθεια. Το θέμα είναι πώς θα χρησιμοποιηθούν τα έσοδα αυτά. Σε μια περίοδο λιτότητας, ε, όταν υπάρχουν νέα έσοδα, όλοι τα θέλουν. Οπότε πρέπει εμείς, στον, αναπτυξιακό τομέα, πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Πρέπει δηλαδή να πούμε ποιοι είναι οι ηγέτε, ποιοι είναι αυτοί που πρωτοστατούν σε αυτή τη διαδικασία και πώ μπορούμε να του κινητοποιήσουμε. Αυτό νομίζω ότι είναι ένα βασικό ε, ζήτημα. Και γι' αυτό νομίζω ότι οι πολίτες και οι ε, σχετικές οργανώσεις πρέπει να ε, εξετάσουν πώς μπορούν να απορροφηθούν τα έσοδα αυτά. Γιατί πολλές φορές έχουμε πει ότι κάτι δεν ήταν δυνατό, τελικά κατέστη δυνατό, γιατί πιο πριν ε, δεν ήταν δυνατό επειδή δεν υπήρχε η απαραίτητη ηγεσία, ούτε ήταν η κατάλληλη στιγμή. Πρέπει λοιπόν κάποιος να εντοπίσει τους πρωτοστάτες προκειμένου να αξιοποιηθούν σωστά και από αναπτυξιακής απόψεως τα επιπλέον αυτά έσοδα. Αυτή είναι η δική μου άποψη για το φόρο χρηματοοικονομικών συναλλαγών. Όσον αφορά την λογοδοσία, Εγώ γνώρισα και τον Πρωθυπουργό και τον Υπουργό Εξωτερικών του Πακιστάν ε, και αυτό ήταν το πρώτο πράγμα που τους είπα. Οι πολίτες μας είναι μεν γενναιόδοροι, αλλά περνούν και αυτή η κρίση. Στις δικές τους χώρες. Και αν θέλετε αυτή η γενναιοδορία να συνεχίσει, ένας μόνος τρόπος υπάρχει. Και αυτός είναι η λογοδοσία. Είχα μάλιστα και μια καλή συζήτηση με τον Πρωθυπουργό του Πακιστάν, για το θέμα αυτό και τώρα μάλιστα υπάρχει πρόταση να υπάρξει μια εθνική ομάδα για την εξασφάλιση της λογοδοσίας. Είναι, ένα, είναι, είναι σχόλια που ακούω πολύ συχνά και ε, στο Κοινοβούλιο, αλλά και από τους πολίτες τους ίδιους. Και να σας πω την αλήθεια με βρίσκει και εμένα σύμφωνη. Ε, και βέβαια δεν, ε, είναι και για μένα πολύ εύκολο πολλές φορές όταν με στριμώχνουν να πω «Α, δεν φταίω εγώ». Ε, με πιέζουν είτε από το Κοινοβούλιο, είτε οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και η μητέρα μου πληρώνει φόρους. Ενδεχομένως ένα σέντ του ευρώ να πηγαίνει στο Πακιστάν. Οπότε και εγώ είμαι υπεύθυνη για αυτό το ένα σέντ που πληρώνει ο κάθε πολίτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, όταν ε, συζητώ με το Πακιστάν ή με άλλες χώρες. Πρέπει λοιπόν να τους εξηγώ κάθε φορά ότι δεν είναι απλώς πλούσιοι άνθρωποι που δεν ξέρουν τι να κάνουν τα λεφτά τους και θέλουν να τα πετάξουν σε μαύρες τρύπες. Υπάρχουν άνθρωποι και άνεργοι, συνταξιούχοι, που και εκείνοι συνεισφέρουν τον οβολό τους. Οπότε κάθε φορά του το λέω και θα συνεχίσω να το κάνω. Αυτό για το θέμα του Πακιστάν. Για τον προπολογισμό τη ε, ανθρωπιστική βοήθεια, ε, εγώ κοιμάμαι ήσυχη γιατί ήρθα σε επαφή με του ε, συνεταίρου μα, γνωρίζω του μηχανισμού που χρησιμοποιούμε. Ένα τρίτο των προγραμμάτων και ένα τρίτο των, του προπολογισμού μας ελέγχεται κάθε χρόνο. Έχουμε και επιτόπου προσωπικό που αξιολογεί την κατάσταση και έρχεται σε επαφή με την τοπική κοινωνία. Όμως εμείς ε, παρέχουμε βοήθεια και όχι ρευστό. Και αυτό κάνει τη δουλειά μας λίγο ευκολότερη. Όμως, δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν και κίνδυνοι. Δηλαδή δεν υπάρχουν κίνδυνοι καταχρήσεων, για παράδειγμα. Οπότε προσπαθούμε να εξασφαλίσουμε ότι γίνεται καλή δουλειά. Πρέπει όμως να προσπαθήσουμε ακόμη περισσότερο γιατί βρισκόμαστε σε δύσκολους καιρούς, ε, περνούμε δύσκολες καταστάσεις και η, η ανθρωπιστική βοήθεια, η ανάγκη ανθρωπιστικής βοήθειας μόνο αυξάνεται. Τώρα, όσον αφορά την ασφάλεια του προσωπικού, του προσωπικού μας. Κοιτάξτε, αυτό με ανησυχεί, δεν κοιμάμαι τόσο ήσυχη για αυτό το θέμα. Πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να βελτιώσουμε την ασφάλειά τους. Μερικές φορές μάλιστα επιδεινώνεται η κατάσταση. Τι να κάνουμε να στείλουμε στρατιωτικέ δυνάμει μερικέ φορέ χρειάζεται. Για παράδειγμα, στη Σομαλία χρειάστηκε με το θέμα τη πειρατεία, αλλά. Είναι δύσκολο κι αυτό. Χάνονται ζωές, γίνονται απαγωγές. Πολλές φορές, ε, όταν έρχομαι σε επαφή με τους ανθρώπους αυτούς, ζητούν μεγαλύτερη ασφάλεια. Πολλές φορές μου λένε, μα πότε θα φύγουμε από εδώ. Και με ρωτούν αν υπάρχουν αποφάσεις σχετικά με αυτό. Για παράδειγμα από τον Ταρφούρ. Λίγο πριν φύγουν δύο ε, μέλη της ε, αποστολής, της ανθρωπιστικής, ήταν θύματα απαγωγής. Πρέπει λοιπόν με κάποιο τρόπο να συνδυάσουμε την ανθρωπιστική βοήθεια και με την εξωτερική πολιτική και να είμαστε και πολύ προσεκτικοί γιατί πολύ συχνά οι άνθρωποι αυτοί θεωρούν ότι η απλούστερη λύση είναι να στείλουμε για παράδειγμα στρατεύματα γιατί θεωρούν ότι είναι ο καλύτερος τρόπος να εξασφαλιστεί η ασφαλειά τους. Και συνεπώς προσπαθώ να σας πω το σύνορα ότι δεν έχω μια πάρα πολύ καλή απάντηση για το πρόβλημα που θέσατε. Όσον αφορά ε, το Ταμείο Ταχείας Αντίδρασης και Αλληλεγγύης, έχουμε ενσωματώσει την ανθρωπιστική βοήθεια στο θέμα της ταχείας ε, ανταπόκρισης. αν υπάρξει ένα πρόβλημα στην Μολδαβία, μπορούμε την επόμενη μέρα να εκταμιεύσουμε 3 εκατομμύρια ευρώ. Αν συμβεί όμως στη Ρουμανία, είναι διαφορετικά τα πράγματα. Μπορεί δηλαδή να καθυστερήσει η αντίστοιχη βοήθεια. Τρει, πέντε, οχτώ μήνες. Και όταν συζητούμε το Ταμείο Αλληλεγγύη, ίσως θα έπρεπε να επιμείνουμε στην ευελιξία, να είναι ένα κίνητρο ετοιμότητας. δηλαδή τα χρήματα να αξιοποιηθούν στον τομέα της ετοιμότητας. Τα κράτη-μέλη όμως μου λένε ότι δεν θέλουν να ξανασυζητηθεί αυτό. Και ο λόγος είναι ότι δεν είναι οι υπεύθυνοι για την ανταπόκριση σε περίπτωση καταστροφών, είναι οι Υπουργοί Οικονομικών που αποφασίζουν. ή, θε, ας πούμε θέλουν να υπάρξει μία ρήτρα αν δεν χρησιμοποιηθεί το Ταμείο Αλληλεγγύης να επιστραφούν τα χρήματα. Εν πάση περιπτώσει θέλω να πω ότι υπάρχουν πολλοί ενδιασμοί Δηλαδή, γιατί δεν μπορούμε να πούμε ότι θα διαθέσουμε 5 εκατομμύρια ευρώ, είτε είναι φτωχή χώρα, είτε δεν είναι φτωχή, σε περίπτωση που υπάρχει μια μεγάλη θεομηνία, για παράδειγμα. Εγώ θα προτιμούσα αυτή τη λογική προσωπικά. Αλλά δεν είμαι πάρα πολύ σίγουρη ότι μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο σε επίπεδο, σε μια περίοδο λιτότητας. Γιατί οι Υπουργοί Οικονομικών σε 23 γλώσσες θα μας πούνε όχι, nine, no, yet. Και το καταλαβαίνω, εντάξει, και εκείνοι τη δουλειά τους κάνουν, πρέπει να προσέχουν τους προπολογισμού τους. Ευχαριστούμε πολύ κυρία Επιτροπέ. Ευχαριστούμε πολύ που ήρθατε μία ακόμη φορά να μας δείτε. μα κάνατε έναν απολογισμό της τεράστιας, ε, του τεράστιου καθήκοντος που φέρατε εις πέρας, με ιδιαίτερη ενέργεια. Σας θαυμάζουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που, μας, ε, που μοιραστήκατε μαζί, μαζί μας το όραμά σας και την ε, το πώς βλέπετε το μέλλον. Ευχαριστούμε πολύ. Υπό τα διάφορα θα ήθελα να σας πω ότι σήμερα το απόγευμα στις 3 η ώρα υπάρχει μια συνεδρίαση στην αίθουσα 4Q2 κοινή μεταξύ Εξωτερικής, ε, Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων και Δικαιωμάτων του Ανθρώπου για την παρουσίαση των ε, υποψηφίων για το γραφείο Ζαχάροφων. Η επόμενη συνεδρίαση θα γίνει στις Βρυξέλλες 25 Οκτωβρίου από τις 3 ε, ως τις 6.30 και την Τρίτη, την επομένη, από τις 9 ως τις 12.30. Πέρα στη συνεδρίαση.